νόμισμα ε, τη Λύρα στην Ιρλανδία για να λύσουμε τα προβλήματα και να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα σοβαρά με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ως Ιρλανδός βουλευτής καθόλου δεν χαίρομαι